Okay, colleague. We just start. Uh, I submit to you the... Σχίζουμε, συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος. Σας υποβάλλω προς έγκριση την εμείς διάταξη και έχουμε ένα νέο σημείο 7 σε σχέση με την ε, ε, έκθεση Κόλλιο για τη λειτουργία της συνθήκης Έγκεν. Αυτό θα γίνει στις 11 και 4. Να λάβετε υπόψη ότι δυστυχώς σε κροατικά και Ιρλανδικά, Κελτικά το στόμα δεν θα έχουμε σήμερα. Αγαπητοί συνάδελφοι και τώρα έχουμε το σημείο ανταλλαγή απόψεων με τον Rob Βουέινραιτ, τον εκτελεστικό διευθυντή της Europol. Πριν από λίγες εβδομάδες συνάδελφοι είχαμε την ακρόαση με την κυρία Ντεμπόλε, την υποψήφιο που θα διαδεχθεί τον κύριο Βουέινραιτ, αλλά σήμερα ε, θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια ε, ανασκόπηση της εννεαετίας κατά την οποία ο κύριος Ράιτ ήταν επικεφαλής της Europol και τον ευχαριστώ για την ε, αφοσίωση στο έργο του, για τον επαγγελματισμό με τον οποίο κράτησε το πιδάλιο από το 9 που ανέλαβε. Η εντολή του θα περατωθεί στις 30 του 18. Uh, first, Mr. Uh, Wainwright will make a presentation, which will be followed by... Είναι μια παρουσίαση και στη συνέχεια ανταλλαγή απόψεων με τους βουλευτές. Κύριε Wainwright, έχετε τον λόγο. Thank you, Madam Chair. Uh, good morning, everyone. Καλημέρα σε όλους, τον κύριο Wainwright. Και χαίρομαι που ήρθα εδώ για τελευταία φορά να σας παρουσιάσω τι έγινε, όπως τόσες φορές άλλωστε έχουμε πει τελευταία εννέα και ίσως το πιο σημαντικό πρόβλημα σήμερα είναι ότι θα πρέπει να σας ευχαριστήσω για την ε, συνεργασία. Τη συνεργασία την θετική που είχαμε ως ε, Europol. Προσπαθήσαμε σε αυτή την περίοδο και πρέπει να σας ευχαριστήσω και για τη δική σας αφοσίωση, για τη δική σας βοήθεια που βοηθήσαμε τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν ε, τους, πολίτε πολίτες της Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευράς και τώρα να δούμε δύο πραγματάκια για αυτή την περίοδο κατά την οποία είχαν λάβει αυτά τα καθήκοντα επικεφαλής της Europol και όπως πολλές φορές τα έχουμε πει στην Επιτροπή σας έχουμε ε, όλο ένα και πιο περίπλοκες απειλές όλο ένα και πιο σημαντικές απειλές στην Ένωση έχουμε βέβαια τα αποτρόπια γεγονότα λόγω τρομοκρατίας τελευταία τριετία, τετραετία πρόκειται για μια τάση που άλλαξαν το πρόσωπο της τρομοκρατίας και ιστορικά αν το εξετάσουμε ως θέμα εθνικής ασφαλείας αλλά και σήμερα είναι θέμα συλλογικής ασφαλείας και αυτό σας το λέω γιατί πια δεν είναι θέμα εθνικισμού, δεν είναι απειλή για την αγκαιρότητα μιας χώρας αλλά το θέμα είναι ο τζιχαντισμός ο διεθνής που έχει διασυνοριακές δυνατότητες. Χρησιμοποιείται η τεχνολογία ε, σαν μια έκφραση της παγκοσμιοποίησης για αυτό το ε, χαλιφάτο. Και έχουμε όλους αυτούς τους ριζοσπαστικοποιημένους Ευρωπαίους οι οποίοι πηγαίνουν και έρχονται από Συρία και Ιράκ. Οπότε και το φαινόμενο είναι πραγματικά διεθνές όσο απειλή στην ασφάλεια. Και όλοι εμείς που ασχολούμαστε εδώ στα θεσμικά όργανα με την ασφάλεια ε, καταλήγουμε στο ότι χρειάζεται συλλογική αντίδραση. Επίσης, θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν διάφορες μορφές οργανωμένου κλίματος και κυβερνών κλίματος. Υπάρχουν ε, πάρα πολλές ε, κινήσεις ε, εμπορία, εντάθηκε αυτό από το 2015. Έχουμε εμπορία ανθρώπων που κατά τη θητεία μου αυτά τα 9 χρόνια ε, πολύ βαθμία και πολύ αργά ξύπνησαν τα κράτη-μέλη για να το αντιμετωπίσουν. Και ακόμα και σήμερα δεν έχουμε στρέψει την προσωπική μας όσο θα έπρεπε και έχουμε χιλιάδες θύματα αυτής της σωματεμπορίας, της εμπορίας ανθρώπων, γιατί τα δύο τρίτα τους είναι ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης που υφίστανται αυτή την ε, σωματεμπορία, αυτή την ελευθερία ανθρώπων. Και έχουμε επίσης και τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Είναι ευάλωτοι και τους εκμεταλλεύονται αυτές οι συμμορίες. Αυτό είναι κάτι σύμφυτο με το μεταναστευτικό και ξέρω ότι σας ενδιαφέρει ιδιαίτερος ως Επιτροπή. Επίσης, σε αυτή την ε, περίοδο είδαμε απάντες μεγάλης κλίμακας, ούτε αυτές τις πρόσεξαμε αρκετά, αλλά η οικονομία πλήγει σε μεγάλο βαθμό. Ήταν ζητήματα ε, εγκλημάτων εις βάρος πραγματικής ιδιοκτησίας και φτάσαμε στα 85 δις ευρώ ετησίως ως ζημία. Και αυτό βέβαια ήταν χτύπημα στην καινοτομία, στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Και αυτό δείχνει το ότι έχουμε αυτές τις επαγγελματικέ μαφίες που εξελίχθηκαν και σε πολλές χώρες και σε πολλούς τομείς της εγκληματικότητας δρούν. Και έχουμε βέβαια συγκέντρωσή τους σε κάποιες χώρες, αλλά πέραν αυτών είναι πάρα πολύ εφευρετικά αυτά τα συνδικάτα του εγκλήματος και βέβαια βοηθούνται από το σκοτεινό ίντερνετ, και τεχνολογία. Μα... Κάποιος πραγματικά επαγγελματίας εγκληματίωση οι οποίοι που έχουν αναλάβει αυτή την, τον τρόπο λειτουργίας και το έγκλημα είναι ε, από τις απειλές που έχουμε με ίσως η πιο μεγάλη δεν έχει τέτοιο αντίκτυπο όπως η τρομοκρατία. Αλλά το πρόβλημα είναι μακροπρόθεσμο γιατί αυτοί οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται τις νέες τεχνολογίες όπως το Darknet, όπως την ε, κρυπτογράφηση, την κωδικοποίηση, όπως αυτά τα κρυπτονομίσματα και είχα επίσης και τις ε, επιθέσεις ιών κατά των υπολογιστών, κατά τις πληροφορικής και στο παρελθόν επίσης είδαμε αυτά τα ψεύτικα email τα οποία πέτυχαν το στόχο τους και αυτό τώρα έχει βελτιωθεί όσον αφορά τα αποτελέσματά τους και τους έχει αποδώσει κέρδη. Και φυσικά ο στόχος ε, είναι τράπεζες κάποιοι πλούσιοι, κάποια θεσμικά όργανα και έτσι έχουμε αυτές τις επιθέσεις που ονομάζονται malware με τους ιούς. Και τελικά αυτό το κυβερνόγκλημα έχει αποκτήσει βιομηχανικό χαρακτήρα. Είναι πολλές χιλιάδες αυτοί που συμμαχούν για να πετύχουν το στόχο τους διάφορα φόρουμ ε, και σε αυτά γίνονται συναλλαγές από ναρκωτικά και όπλα μέχρι υπηρεσίες σεξ και είναι μεγάλη απειλή αυτή η οργανωμένη δραστηριότητα. Και επίσης κάτι άλλο που έχει ανθεί τελευταίο 1,5 χρόνο. Έχουμε σύγκληση αυτών των δραστηριοτήτων ε, και που πολλές φορές έχουν ε, χαρακτήρα οργανωμένου εγκλήματος και σχετίζονται πολλές φορές με κράτη. Έτσι αναβαθμίζονται ο πλευράς δυνατοτήτων, ο πλευράς καινοτομίας, οπότε και οι πιο προστατευμένοι είναι πλέον ευάλωτοι σε τέτοιες επιθέσεις. Όλα αυτά είναι η σημερινή τάση του εγκλήματος όλα αυτά πιο διεθνεί, σε πιο μεγάλη κλίμακα, πιο περίπλοκα και οπωσδήποτε έτσι έχουμε για την Europol ε, πιο βαριές ευθύνες. Βεβαίω αντιδράσαμε πρώτα με την βοήθεια του θεσμικού πλαισίου της Ένωσης να είμαστε σαφείς δηλαδή. Ο τρόπος με τον οποίο ο νομοθέτης ε, προέβλεψε ισχυρότερους ε, κανονισμούς και οδηγίες για να ελέγξουμε τα ταξίδια των τρομοκρατών ε, προσφάτως, κάτι το οποίο περιόρισε κατά πολύ την ροή ξένων μαχητών ε, στην Συρία και το Ιράκ. Ε, συνεχίζουμε δε να επεξεργαζόμαστε την οδηγία ξεπλήματος του χρήματος. Έχουμε λοιπόν μια ρυθμιστική αντίδραση και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει αντίκτυπο. Βεβαίω, όσον αφορά την Europol, Επί των ημερών μου είχαμε δύο αλλαγές στο νομικό πλαίσιο. Πιο πρόσφατο ήταν η έγκριση του κανονισμού της Europol το 2017, ένας κανονισμός που επηρεάστηκε πολύ από την Επιτροπή αυτή με πολύ επικοδομητικό τρόπο. Οι πόροι που έχουμε λάβει από τον προϋπολογισμό έχουν διπλασιαστεί σήμερα. Είμαστε 1200 άτομα στη Χάγη και ο προπολογισμό διπλασιάστηκε. Έχουμε ένα προπολογισμό 22 εκατομμυρίων. Ο ρόλος ε, των ε, κρατών μελών επίσης αφορά την στήριξη ε, των τρίτων χωρών. Χωρίς τη δικιά τους την πείρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και βασιζόμαστε στο ότι διασυνδέουμε μια μεγάλη κοινότητα τέτοιων υπηρεσιών. Και η εμπιστοσύνη που έχει αναπτυχθεί φαίνεται στο ότι την περίοδο αυτή οι σύνδεσμοι στην Europol πλέον έχουν αυξηθεί σε 220 άτομα που εκπροσωπούν τις εθνικές τους αρχές από 40 χώρες. Πουθενά αλλού στον κόσμο δεν υπάρχει τόσο μεγάλη συγκέντρωση διοκτικών αρχών και αυτό ακριβώς ε, ενισχύει τις δυνατότητες της Europol να καταπολεμήσει το έγκλημα και την τρομοκρατία. Και βασικό θέμα στο πώς μπορούμε να κάνουμε δουλειά μα είναι τα κέντρα αριστείας, όπως ε, παραδείγματο χάρη το κέντρο κυβερνοεγκλήματος που θεωρείται σήμερα από τα κορυφαία διεθνώς. Το κέντρο παράνομη μετανάστευσης ε, που αυτή τη στιγμή αριθμεί ε, πάνω από 100.000 άτομα έχουμε βρει 17.000 υπόπτους ήδη και βέβαια στο κέντρο αντιτρομοκρατίας όλα αυτά συνέβησαν επί των ημερών ακριβώς για να εστιάσουμε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο την, ε, και να συγκεντρώσουμε την εμπειρία των ευρωπαϊκών Διεκτικών αρχών σε αυτούς τους τομείς ε, προτεραιότητας. Το, για το κέντρο αντιτρομοκρατίας Έχουμε συζητήσει και εδώ και αλλού το θέμα του πώς μοιραζόμαστε τις ε, πληροφορίες. Ήταν πρόκληση να πείσουμε τις υπηρεσίες ασφαλείας να δώσουν περισσότερα δεδομένα στην Europol. Και αυτό συνέβη τα τελευταία δύο χρόνια. Το σύστημα πληροφοριών λοιπόν της Europol έχει αυξήσει τον αριθμό των πληροφοριών που λαμβάνει από τα κράτη-μέλη. Πριν από δύο χρόνια είχαμε γύρω στις 2.000 σχετικές εκθέσεις που αφορούσαν την τρομοκρατία στο σύστημά μας. Σήμερα είναι 500.000 σε δύο χρόνια. Και αυτό δείχνει το ότι τα κράτη-μέλη μοιράζονται περισσότερες πληροφορίες. Επίσης, ε, πέρσι υποστηρίξαμε 439 επιχειρήσεις ε, σε σχέση με 227 το προηγούμενο έτος και αυτό ακριβώ δείχνει την ίδια τάση. Και σε γενικές γραμμές ε, τα εννέα χρόνια της ε, θητείας μου υπήρξε έννοια πλασιασμός των διασυνοριακών υποθέσεων που στηρίζουμε. Οπότε υπάρχει και αυτή η αύξηση του φόρτου εργασίας ε, καθώς η ζήτηση αντιμετωπίστηκε με περισσότερη προσφορά από μέρου μας και προσπαθούμε να διαχειριστούμε τον όγκο των πληροφοριών. Βεβαίως έχουμε, όπως είπαμε, 1.200 άτομα και ακριβώς έχουμε ένα μοναδικό εύρος όσον αφορά τις ε, υπηρεσίες, ε, τις διάφορες διοκτικές αρχές και θα έλεγα ότι έχουμε το πιο προχωρημένο μοντέλο Προστασία δεδομένων από ανάλογε υπηρεσίε στον κόσμο και έτσι έχουμε την εμπιστοσύνη, την αυτοπεποίθηση να συλλέγουμε δεδομένα σε τόσο μεγάλη κλίμακα και με ένα πλαίσιο προστασία δεδομένων ώστε να είμαστε αξιόπιστοι, να συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα που χρειαζόμαστε, να διακρατούμε μόνο τα δεδομένα που χρειαζόμαστε, πάντα αναλογικά με τον σκοπό, την καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Νομίζω ότι έχουμε αναπτύξει πολύ σύγχρονες ε, δυνατότητες ε, ανάλυσης δεδομένων για να μπορούμε να διαχειριστούμε τις τεράστιες ποσότητες δεδομένων που λαμβάνουμε. Το 2017 για πρώτη φορά περάσαμε το όριο του ενός εκατομμυρίου μήνυμάτων που ανταλλάχθηκαν σε ένα έτος στο δίκτυο της Europol ε, και πλέον αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο φόρτο εργασία, αλλά είναι και η δουλειά μας και η ανάλυση ακριβώς μας επιτρέπει να δούμε την διασυνοριακή διάσταση του εγκλήματο και της τρομοκρατίας. Σημαίνει λοιπόν πως ε, όλα αυτά μας έχουν δώσει την ευκαιρία να έχουμε αποτελέσματα και να επηρεάσουμε το έγκλημα και την τρομοκρατία. Το επίπεδο εμπιστοσύνη έχει ανέβει. Σύμφωνα με την έρευνα των εταίρων μας βλέπουμε ότι η ικανοποίηση είναι 72% το υψηλότερο επίπεδο που είχαμε ποτέ σε σχέση με 57% πριν από 10 χρόνια. Ελπίζω επίσης ε, σε συνεργασία με την Επιτροπή μας ότι μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε την γνώση μας και την επιρροή μας για να διαμορφώσουμε το πώς ε, αναπτύσσεται η νομοθεσία και η πολιτική. Γιατί το νομοθετικό περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργούμε θα πρέπει να επηρεάζεται και από την δική μας ε, την γνώμη ως εμπειρογνώμονες. Ε, υπάρχουν βεβαίως πολλές απογοητεύσεις που σχετίζονται με το έργο μας ε, και θα ήταν παράληψη να μην αναφέρω τους ε, πόρους όχι μόνο της Europol αλλά συνολικά των ε, υπηρεσιών εκείνων που προσπαθούν να διατηρήσουν την εσωτερική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι συνολικά είναι χαμηλά τα ποσά και αναντίστοιχα με την απειλή. Θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμα σοβαρά παραδείγματα συστημικής αδράνειας ε, στην ε, προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε κάποια από αυτά τα περίπλοκα προβλήματα. Χαρακτηριστικό του τους mm. έχουμε την οδηγία περί ξεπλήματος χρήματος που είναι εντυπωσιακά αναποτελεσματική στο να κάνει την δουλειά μας. Ε, ε, πρόκειται για μια τεράστια επένδυση που κοστίζει και δισεκατομμύρια και στις τράπεζες, οπότε ε, δεν είναι τόσο εύκολο να τις κατηγορήσουμε. Απλά έχουμε σχεδιάσει ένα σύστημα τα τελευταία χρόνια, το οποίο είναι τελικά αναποτελεσματικό, παροχημένο και συγκεκριμένα δεν υπάρχει η δυνατότητα να βρεθούν τις πληροφορίες αυτοί που τις χρειάζονται. Και νομίζω πως μια σοβαρή αναθεώρηση αυτού του πλαισίου απαιτείται αν είναι ε, να λέμε στα σοβαρά ότι ακολουθούμε το χρήμα γιατί δεν το κάνουμε αυτή τη στιγμή και ακριβώς δίνει την δυνατότητα στο έγκλημα να ανθεί. Τέλος, να ευχαριστήσω και πάλι τον ρόλο του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σας ιδιαίτερα ε, όσον αφορά τις ε, πρακτικές πτυχές ε, του προϋπολογισμού, των πόρων και το να ακούγεται τη φωνή μας στην σύνταξη της νομοθεσίας. Συχνότερα βεβαίως μας ακούει το Κοινοβούλιο παρά το Συμβούλιο. Για το γνωρίζουμε αυτό και το αναγνωρίζω και είμαι ευγνώμων. Επίσης το γεγονό ότι έχετε κάποιες ε, εξειδικευμένες επιτροπές που ασχολούνται με το θέμα προληπτικά, όπω η Επιτροπή για την Τρομοκρατία. Έχουμε όλο και σχέση λοιπόν με το Κοινοβούλιο, όχι μόνο γιατί είναι μια ρυθμιστική και θεσμική απέτηση, αλλά μας ε, δίνει περισσότερη, σημαίνει περισσότερη λογοδοσία και άρα περισσότερη αξιοπιστία με το, προς το κοινό, την κοινή γνώμη. Και να σας ευχαριστήσω και πάλι προσωπικά και τους οπόντες ε, και την Επιτροπή σας. Ε, δεν ε, συμφωνούσαμε πάντα. Έτσι είναι τα πράγματα στην δημοκρατία. Αλλά προσπάθησα να υπηρετήσω σωστά τα καθήκοντα που μου ανατέθηκαν και ένα λογοδοτό ενώπιον του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την ε, πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία σας ευχαριστούμε κύριε Βαϊνράιτ. Έχω εγώ ένα ερώτημα, κύριε Βαϊνράιτ. Μπορείτε να μας πείτε κατά τη γνώμη σας τι είδους όχι, να το πω αλλιώ. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερε επιτυχίε σα κατά την εννέα θητεία σας. Και ποια και τι είδους προβλήματα αντιμετωπίσατε με κάποιες δραστηριότητες, κάποιες ιδέες που ενδεχομένως είχατε και δεν μπορέσατε να ε, υλοποιήσατε μέχρι σήμερα. Θα δώσω το λόγο τώρα στους ε, συναδέλφους, πρώτα στους συντονιστές. κυρία Ζήπελ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη που άργησα. Παρ' όλα αυτά, όταν μιλήσατε για το hacking, μου δώσετε την ευκαιρία να θέσω ένα θέμα που συζητήσαμε και πρόσφατα στη συνεδρίαση των συντονιστών τη Δευτέρα. Θα θυμάστε ότι το 2013 υπήρχαν κατηγορίες ότι υπήρξε χακάρισμα των υπηρεσιών της Belgacom από μυστικές υπηρεσίες και είχαμε μάλιστα σε συνεδρίαση ε, απευθύνει ερωτήματα στην Belgacom, στους υπεύθυνους προστασίας προσωπικών δεδομένων ε, Belgacom ε, και σε εσάς. Σε εκείνη την ακρόαση είχατε πει ότι δεν είχατε λάβει αίτημα για να διερευνήσετε αυτό το χακάρισμα. Ωστόσο πριν από λίγες εβδομάδες ε, δημοσιεύθηκε ότι υπήρξε τελικά αίτημα των βελγικών αρχών προς την ε, Europol και ε, ακριβώς ε, ο ρόλος σας είναι να εξασφαλίζετε την ασφάλεια και στις τηλεπικοινωνίες. Φαίνεται όμως ότι αρνηθήκατε να ερευνήσετε και να παρέχετε την συνδρομή σας σε αυτή την υπόθεση. Μπορείτε να μας εξηγήσετε άλλη μια φορά γιατί η Europol αρνήθηκε να βοηθήσει το Βέλγιο στη συγκεκριμένη έρευνα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Έρνστ. Ο, δεν περίμενα να μου δώσετε τόσο γρήγορα το χρόνο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα εκ μέρους της ΓΚΟΕ να σας ευχαριστήσω κύριε Βάινράιτ. Ήταν πραγματικά ε, δύσκολες συζητήσεις που είχαμε πολλές φορές. Ε, ε πηγάζει από τη φύση των ε, πραγμάτων αυτό βεβαίω. Αυτό βεβαίω δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει η Europol να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο για τη δικτύωση των αστυνομικών αρχών για την διαρθρωμένη ε, συνεργασία, ιδιαίτερα στον τομέα τη τρομοκρατία. Αυτό προφανώ είναι αναμφισβήτητο. Υπήρχαν πολλές, ε, πολλά περιστατικά τα τελευταία χρόνια που αποδεικνύουν ότι ακριβώ η συνεργασία των αστυνομικών αρχών, η δικτύωση αυτών και η ανταλλαγή πληροφοριών, η ροή των πληροφοριών ε, δεν υπήρξε απρόσκοπτη, να το πω έτσι. Φυσικά εμείς ε, το επικρίναμε αυτό το, το φαινόμενο ως πολιτικά, πολιτική ομάδα πάντοτε. Όμως στο θέμα της τρομοκρατίας πρέπει κανείς να λαμβάνει υπόψη του πάρα πολλούς παράγοντε και πάρα πολλά στοιχεία. Είναι περίπλοκο το ζήτημα, αλλά πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα στην πρόληψη, όχι ως μαϊντανό, γιατί πάντα πρέπει να μιλάμε και για την πρόληψη σε όλα τα θέματα, στα σοβαρά και ε, να συζητήσουμε πώ ακριβώ θα καταπολεμήσουμε τα γενεσιουργά αίτια. Και αυτό βεβαίω δεν αφορά ως ε, ε, αρμοδιότητα αποκλειστικά τη Europol, προφανώ και όχι, είναι ένα γενικό, γενικό καθήκον τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρώ ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν γίνει επαρκείς προσπάθειες, διότι γνωρίζετε ότι η τρομοκρατία είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να το λύσει κανεί μόνο αστυνομικά. Το άλλο θέμα είναι ότι υπάρχει, χρειάζεται μια ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την εξασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γνωρίζετε ε, ότι ω Κοινοβούλιο ε, μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ ε, αυτό το ζήτημα της ισορροπίας μεταξύ ασφάλειας και τήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γι' αυτό και ζητούμε πάντοτε ως ε, Κοινοβούλιο για τη διαφάνεια. Ε, είχαμε και στο σχετικό κανονισμό, στις συζητήσεις που είχαν γίνει για, το για τον λόγο κανονισμό, είχαμε ε, δραστηριοποιηθεί αυτό. Χρειαζόμαστε ένα ενερμονισμένο σύστημα προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ευρώπη. Προφανώς τα δεδομένα που επεξεργάζεται η Europol δεν είναι δεδομένα εξωγήινων, είναι Ευρωπαίων πολιτών και γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε ε, έναν σαφή ορισμό και έναν σαφή κατάλογο αρμοδιοτήτων και κριτηρίων με τα οποία θα επεξεργάζεται η Europol τα δεδομένα. Είναι ένα θέμα κανθόδες προφανώς. Παρ' όλα αυτά πρέπει να, καταλήξουμε, θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμβασμό. Εμείς ως εισηγήτρια σας το λέω θα απαλέψουμε, ε, θα αγωνιστούμε για αυτό το θέμα Βεβαίω πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε λύση. Η λύση αυτή όμω δεν μπορεί να είναι να πούμε ότι δεν θα κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό και σα ε, το λέω με την ευκαιρία τη παρουσία σα σήμερα εδώ για να μπορείτε να διαβάσετε και στου συναδέλφου σα το μήνυμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ ο κύριο Λένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Wainwright που είστε εδώ και για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε τα τελευταία χρόνια ε, με την Επιτροπή μας και για τις προσωπικές σας προσπάθειες που καταβάλλετε για να αυξηθεί η ασφάλεια των πολιτών. Το εκτιμούμε αυτό και ως πολιτική ομάδα. Εσείς ε, ευχαριστήσατε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σας ευχαριστούμε που μας ευχαριστείτε για το ότι ε, σας εξασφαλίσαμε τον προπολογισμό που χρειάζεται. Όμως είπατε ότι τα χρήματα που διατίθεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ λίγα σε σχέση με την με το μέγεθος και την κλίμακα των απειλών που αντιμετωπίζουμε. Πώς πιστεύετε δηλαδή πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα, τι παραπάνω πρέπει να δώσουμε, πρέπει να δώσουμε περισσότερους πόρους, ε, πώς μπορούμε καλύτερα να προετοιμαστούμε ε, απέναντι στις απειλές που αντιμετωπίζουμε. Επίσης, είπατε για τον πλούτο επιλοφοριών που έχει στις βάσεις δεδομένων της Europol. Γνωρίζετε ότι στο Κοινοβούλιο ε, επεξεργαζόμαστε το ζήτημα της διαλειτουργικότητας με τα κεντρικά ευρωπαϊκά συστήματα και τα δεδομένα της Ευρωπόλ με κάποιον τρόπο συνδέονται με αυτό το θέμα, αλλά όχι και τελείως. Πώς ε, λοιπόν πιστεύετε ότι οι πληροφορίες που έρχεται ως Europol μπορούν να ε, ωφελήσουν το ζήτημα της ε, διαλειτουργικότητας. Και τέλος, τα 9 χρόνια που, της θητείας σας είχαμε ένα πολύμορφο ε, τοπίο κανονισμών και οδηγιών νομοθετικού πλαισίου δηλαδή ε, και έχετε μεγάλη εμπειρία. Ποιε πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι οι μελλοντικέ νομοθετικέ πρωτοβουλίε, σε ποια ε, κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν. Ευχαριστώ, κυρία ε, Γκροπίν. Thank you very much. <laughs> Okay. În primul rând, uh, vreau să Πρώτα πρώτα ευχαριστώ για την ευθύτητα με την οποία μας ε, παρουσιάσατε τις πεπιθήσεις σας, τις ιδέες σας. Ε, βέβαια και υπάρχουν θέματα τα οποία ακόμη εκκρεμούν, πρέπει να τα διεκπαιρεώσουμε. Ε, είναι φυσικό κάποια να γίνει, κάποια να μην έχουν γίνει και άλλωστε ο κόσμος έχει προσδοκίες από την Europol. Θέλει η Europol να τους εξασφαλίζει, να καθησυχάζονται. Με αυτός είναι ο ρόλος της Europol και μας είπατε ότι ε, τώρα έχει ενταθεί η ριζοσπαστικοποίηση και δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η ασφάλεια μόνο σε εθνικό επίπεδο και θα πρέπει να δράσουμε συλλογικά. Μα τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να αντιδράσουμε έτσι συλλογικά και μας είπατε ότι θα πρέπει να είσαστε σύνδεσμο μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών. Ναι, αυτό θα ήταν το ιδανικό, το ιδιώδες. Αυτό, να είστε ο σύνδεσμος. Και επίσης μας είπατε τα θέματα του προϋπολογισμού, της προϋκοδότησης, μας είπατε για την αδράνεια του συστήματος. Εγώ προέρχομαι τον χώρο των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Για πέστε μας όμως πώς θα ταρακουνήσουμε τα πράγματα ούτως ώστε να σταματήσει αυτή η αδράνεια του δημόσιου τομέα. Και βέβαια για το Συμβούλιο και τη δίκιο για τις τρικλοποδιές που βάζει. Πάντω εμεί τι να κάνουμε για αυτή την αδράνεια. Δεν έχουμε προτάσει. δεν ξέρουμε τι να κάνουμε για να ταρακουνήσουμε το σύστημα. Σταματήσει αυτή η αδράνεια. Και γύρω από και άλλε υπηρεσίε δουλεύουν σε, μέσα σε δίκτυο, ε, άρα θα πρέπει και εδώ να δράσουμε συλλογικά. Α, σήμερα το πρωί μάθαμε για τέσσερι που μαχαιρώθηκαν σε ένα κράτο μέλο. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτό το, οργανωμένο έγκλημα, αλλά και τι ε, απάτε. Νομίζω ότι η κατάσταση έχει ξεπεράσει το οικονομικό επίπεδο στο οποίο μας αναφέρατε, το, το, το κόστος. Επέστε μας τη χρειάζεται και εμείς θα τα πούμε στα άλλα θεσμικά όργανα. Ο κ. Ευχαριστώ. Εντάξει. Λειτουργεί το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ. Επαναλαμβάνω αυτό που έλεγα εκτός μικροφώνου. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, για το έργο σας. Σας εύχομαι ε, ό,τι καλύτερο για το μέλλον και στην Ευρωπόλη να ε, οδηγηθεί σε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Ξέρουμε ότι τα προβλήματα αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια και ότι η κλίμακα και το πρόσωπο, η φύση των προβλημάτων αυτών, του εγκλήματος της τρομοκρατίας ε, ε, έχει αλλάξει. Τα γνωρίζουμε αυτό. Όμως έχουμε φτάσει σε ένα ε, σημείο το οποίο γνωρίζετε αλλά δεν αναφέρατε και που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των μελών της Europol. Δεν αναφέρομαι μόνο σε τεχνική κατάρτιση, αλλά και σε ε, εκπαίδευση σε ζητήματα πολιτικών δικαιωμάτων ή και διανοητική αν θέλετε, εκπαίδευση, γιατί οι νέες προκλήσεις ε, απαιτούν νέους τρόπους αντιμετώπισης, χωρίς βεβαίως να ξεχνούμε την υπεράσπιση, την αναγκαία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είπε και η συνάδελφός μου. Κατά τη γνώμη μου, οι ελευθερίες και η ασφάλεια αποτελούν δύο πολύ σημαντικές αξίες. Δεν βρίσκονται όμως ακριβώς στο, στο ίδιο επίπεδο. Ολοκληρωτικά, στα ολοκληρωτικά καθεστώτα η ασφάλεια είναι ύψης της σημασίας. Κάποιες φορές λοιπόν για να μπορεί κανείς να έχει μεγαλύτερη ασφάλεια ζητά ταυτόχρονα να περιορίζονται οι ελευθερίες. Η ασφάλεια καταπιέζει δηλαδή τις ελευθερίες. Στα δημοκρατικά καθεστώτα η ασφάλεια θα έπρεπε να υπηρετεί τις ελευθερίες. Δεν θα, δεν θα πρέπει να καταστέλει η ασφάλεια τις ελευθερίες, να τις περιορίζει, αλλά αντίθετα να τις προστατεύει και να τις υπερασπίζεται. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει καν, κανείς, ε, μάλλον πρέπει να υλοποιείται από ανθρώπους που τα γνωρίζουν αυτά, που πιστεύουν σε αυτές τις, ε, σε αυτές τις αρχές και θέλουν να τις εφαρμόσουν. Τι, τι, ποια είναι η γνώμη σας λοιπόν για την εκπαίδευση, την παιδεία των ε, μελών της ε, Europol. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσινίτση. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Γουένραιτ, όχι μόνο για την παρουσίασή σας αλλά και για το έργο σας για όσα πέτυχε αυτά τα 10 χρόνια η Europol. Γιατί όπως είδαμε, αναπτύξατε τι δραστηριότητες της Europol και όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά για το τι συγκεκριμένα έκανε η Europol. Και το πιο σημαντικό είναι το ότι διευκολύνανται την ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών. Και βέβαια μπορέσατε, όπως είπατε, διασυνοριακά να δράσετε. Και πάλι σας ε, ευχαριστούμε. Έχουμε πάει επανειλημμένα στη Europol για να ενημερωθούμε. Και όντως διαπιστώσαμε πόσο έχει στρέψει την προσοχή της η υπηρεσία σε συγκεκριμένους εγκληματικούς τομείς και δραστηριότητες. Ακριβώς όπως τα είπατε και εσείς. Και έχουμε και την ε, υπηρεσία και το κυβέρνο έγκλημα τώρα στα οποία δράτε. Αλλά όπως είπατε έχουμε τα χρηματοοικονομικά εγκλήματα που έχουν και αυτά φύση διασυνοριακή. Έχω ξέπλυμα χρήματος, ε, εμβάσματα και πότε θα πρέπει η νομοθεσία να προσαρμοστεί σε αυτά, να επικαιροποιηθεί. και για το ξύλινο χρήματος και όχι μόνο γι' αυτό. Οπότε η Europol ίσως θα έπρεπε να πρικοδοτηθεί ούτως υπήν με μια εξειδικευμένη υπηρεσία που να ασχολείται με αυτά τα χρηματοοικονομικά εγκλήματα. Γιατί πολλές φορές αυτές οι επιλήψιμες ε, συναλλαγές αποσκοπούν στο να χρηματοδοτήσουν την τρομοκρατία. Μας είπατε επίσης για τις μαφιόζικες δραστηριότητες και γενικότερα του οργανωμένου εγκλήματος. Είδαμε τι έγινε με την ανθρωποκτονία του Κούτζακ, του δημοσιογράφου στην Σλοβακία. Και είδαμε βάσει των δημοσιογραφικών πληροφοριών ότι έχει ανακατευτεί η Ιταλική μαφία εκεί. Πάντω, εγώ νομίζω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο λίγα έχουμε κάνει σε αυτό το επίπεδο. Και γι' αυτό και κάθισα και έκανα κάποια έρευνα για να δω και να επισημάνω ακριβώ τώρα να συγκρίνω τι γίνεται σε διάφορε ε, χώρε όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα. Θα πρέπει να βρεθεί και ένα κοινό ορισμό και στη συνέχεια αυτό να οδηγήσει σε καλύτερο νομοθετικό συντονισμό. Και επίσης να σας ε, πω αν και κάτι άλλο. Τι γίνεται για αυτές τις πρόδρομες ουσίες των εκρηκτικών που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες. Εδώ θα πρέπει και νομοθετικά να βελτιωθούμε για να καλύψουμε και αυτήν την δραστηριότητα. Τελευταία, τελευταία μου σκέψη που θέλω να σας απευθύνω. Δουλεύω στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, την Ειδική Επιτροπή κατά της τρομοκρατίας και εκεί συνομιλούμε με διάφορους ε, ειδικού του θέματος και αναδύθηκε ένα θέμα που μας ε, ανησύχησε όπως και ο σύνδεφος μίλησε για πρόληψη ε, και εγώ θέλω να δω τι μπορεί να γίνει για την ε, πρόληψη. Πάνω σε αυτό σας ερωτώ. Τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να παρέμβουμε προληπτικά, θεωρείτε ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Θεωρείτε ότι υπάρχει σενάριο ευρωπαϊκής επίθεσης με χημικά. Ήδη έχουμε τέτοιες απαρχές ενδείξεων για κάτι τέτοιο. Θεωρούμε ναι, αλλά τέλος πάντων εσείς από όσα ξέρετε τι θα μπορούσε να γίνει για να αντιμετωπίσουμε τέτοιο κίνδυνο. And Mrs. Και η κύρια Γκίγιομ. Ευχαριστώ κύριε Μπράβο για τη δουλειά σας όλα αυτά τα χρόνια. Μας ε, είπατε κι εσείς για τις καμιά φορά υπερβολικά ζωηρές συζητήσεις που έχουμε κάνει εδώ. Καλή επιτυχία στα μελλοντικά σας καθήκοντα. Οι συνάδελφοι κάλυψαν πολλά θέματα. Πάντως ε, ήταν σωστό το ότι αναφερθήκατε στο κυβερνό έγκλημα, αναφερθήκατε στην καταπολέμηση του ξεπλήματος. Ε, είναι σαφές ότι... Ε, από την εραστεχνική φάση περάσαμε στην βιομηχανική ούτως επί τα τελευταία χρόνια και μας είπατε για αυτά τα προβλήματα της προκλήσεις που έχει η υπηρεσία ως να αφορά τους εταίρους της γιατί θα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών και Europol. Πώς μπορούν να προχωρήσουν τα πράγματα, να εξελιχθεί η κατάσταση. Μα ε, όπως είπατε και εσείς είναι και θέμα όγκου, ποσότητας πληροφορία. Μιλάμε για εκατομμύρια εγγράφων. Σήμερα έχουμε την επίτηση του 8 Μαρτίου. Για πέστε μας, τι, λέτε για τη μαστροπία, για το δουλεμπόριο, Ε, είναι κάτι αρχαϊκό θα μπορούσε να πει κάνει για το σημερινό κόσμο, αλλά από την άλλη μεριά χρειάζεται ε, έντονη καταπολέμηση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τι ερωτήσει. Τώρα θα ακούσουμε απαντήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Κυρία Πρόεδρε, ρωτήσατε για την μεγαλύτερη επιτυχία που είχαμε. Είχαμε αρκετές επιχειρησιακές επιτυχίες, ε, που είναι βεβαίως επιτυχίες των κρατών μελών. Μία την οποία διευκολύναμε εμείς. Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια μια σημαντική επιχείρηση, που τότε αφορούσε την οποια διευκολυναμε εμεις θυμαμαι πριν απο πολλα χρονια μια σημαντικη επιχειρηση που τοτε φορουσε την αποκαλυψη του μεγαλύτερου δικτύου κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. έτσι <coughs> την διάσταση του θέματος και ε, απέκτησε γεωπολιτική εμπιστοσύνη του κοινού. Και πιο πρόσφατα βεβαίω είχαμε τις επιθέσεις στο Παρίσι το 2015 και η ε, αντίδρασή μας, γιατί ήταν η πρώτη φορά που είχε κληθεί η Europol να παίξει έναν τέτοιο υποστηρικτικό ρόλο σε τρομοκρατικό χτύπημα στην Ευρώπη. Είχαμε επίσημο αίτημα από τον Γάλλο εισαγγελέα και ένα τεράστιο ρόλο στο να βοηθήσουμε τις γαλλικές και τις βελγικές αρχές και πραγματικά άλλαξε τον τρόπο που έβλεπαν την Europol οι αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες που ήταν το τελευταίο οχυρό του, των διεκτικών υπηρεσιών που δεν παίζαμε κάποιον ρόλο. Η μεγαλύτερη επιτυχία νομίζω ήταν η δυνατότητά μας να καταφέρουμε να οργανώσουμε μια κοινότητα 1200 ε, αστυνομικών από διαφορετικούς ε, πολιτισμούς ε, και νομίζω ήταν μια μεγάλη επιτυχία μας. Η κυρία Σίπελ επίσης έκανε ένα ερώτημα. Το θυμάμαι, το έχουμε συζητήσει 2013-2014 γεγονό είναι ότι τότε δεν υπήρχε επίσημο βελγικό αίτημα, δεν αποφεύγω το θέμα. Οι βελγικές αρχές ε, ε, έδωσαν ε, βεβαίως τι λεπτομέρειες της επίθεσης στην πλατφόρμα της Europol και το έστειλαν και σε εμάς το μήνυμα και ζήτουσαν πληροφορίες, αν κάποιος έχει πληροφορίες και κατέστησαν σαφές ότι υποψιάζονταν ότι υπήρχε μία δραστηριότητα με τη στήριξη κάποιου κράτους. Εμείς απαντήσαμε ότι δεν είχαμε κάποιες πληροφορίες και κατέστησαν σαφές ότι ε, αυτό ήταν η αντίληψη του κράτους μέλους και η εντολή μας η νομική ήταν σαφής ότι δεν μπορούσαμε πλέον να κάνουμε κάτι αν υπήρχε αυτή η αντίληψη. Οπότε ειδοποιήσαμε γέρος και μετά δεν συνέβη τίποτα. Και από όσο ξέρω δεν έχει αλλάξει τίποτα σχετικά. Πέρα από αυτό το οποίο αναφέρατε τώρα, ένα ρεπορτάζ ενό δημοσιογράφου, το οποίο είναι ανακριβές, παρά το ότι εμεί ήμασταν ανοιχτοί και δώσαμε όλε τι πληροφορίε για του νομικού περιορισμούς που αντιμετωπίζουμε, αλλά τα παρουσίασε με τρόπο παραπλανητικό. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν προκύψει νέε πληροφορίε. Η συζήτηση τότε, θυμάμαι, με τους ε, συναδέλφους και ένα-δύο μέλη της Επιτροπής, Κατέληξε στο ότι ήταν λυπηρό ότι δεν είναι αυτό μέρος της εντολής μας και βεβαίως ο νομοθέτης είχε τη δυνατότητα να το αλλάξει αυτό, αλλά αποφάσισε να μην το κάνει. Οπότε σήμερα είμαστε στην ίδια θέση όπως ήμασταν τότε και δεν θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ένα τέτοιο αίτημα. Ο κύριος Έρνστ και άλλοι ρώτησαν για τον ε, ρόλο μας στην πρόληψη της τρομοκρατίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, ειδικά στον ψηφιακό χώρο, όπου ακριβώς κάνουμε μεγάλη δουλειά στον τομέα της πρόληψης σε 80 πλατφόρμες κοινωνικών μέσων για να βρούμε ακριβώς ε, τρομοκρατικό περιεχόμενο. Βεβαίως ε, η καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίηση δεν είναι δουλειά μας. Ε, και είχατε βεβαίω δίκιο για την ισορροπία με τα θεμελιώδη δικαιώματα και αναγνωρίζουμε την δουλειά που έχει κάνει η συγγήτρια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και βεβαίως το σκεπτικό του να έχουμε ένα εναρμονισμένο σύστημα και αντιλαμβανόμαστε την σημασία του. Αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι πριν από ένα έτο η Επιτροπή σα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να ε, φτιάξει ένα μέσο προστασία προσωπικών δεδομένων για την Europol. Πολύ σημαντικό. Οπότε έχει αλλάξει το νομικό μας πλαίσιο σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και αυτό παρουσίασε κάποιες πρακτικές και ε, νομικές ε, δυσκολίες. Βέβαια, αν ο στόχο είναι ένα εναρμονισμένο σύστημα, το αντιλαμβανόμαστε, ε, καθώς αρκεί να διατηρούνται τα ωφέλη του να έχουμε, όπως είπαμε, ένα τόσο εξελιγμένο σύστημα προστασίας των δεδομένων. Ο κ. Λένερτ μίλησε για τον προϋπολογισμό. Είχαμε αυξήσει ε, του προϋπολογισμού, αλλά συνολικά ξέρετε ότι το μέγεθο ε, του προπολογισμού για θέματα ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά μικρό. Ε, δεν βγάζω νούμερα έτσι όπως μου έρχονται, είναι αποτέλεσμα εκθέσεων των θεσμικών οργάνων. Η διαλειτουργικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική και βεβαίω εμεί μπορούμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο καθώς μπορούμε με ένα σύστημα προστασία δεδομένων να έχουμε διάφορα συστήματα πληροφοριών. Η κύρια προτεραιότητα βέβαια πρέπει να είναι η κυβερνοασφάλεια. Αλλά σε ένα συγκεκριμένο θέμα θεωρώ ότι ο κανονισμό κατά του χρήματος επίσης πρέπει να εξεταστεί και η κυρία Τσινίτσι μάλιστα ρώτησε αν ε, θα πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο κανονισμό για το ξέπλυμα χρήματος. Επίσης, ε, περιλαμβάνει και την δουλειά που κάνουμε για το δίκτυο FRU. Αλλά βεβαίως ε, κάτι το οποίο μας απογοητεύει είναι ότι η αναθεώρηση της σχετικής οδηγίας είναι ένα απλό βήμα για να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε διεθνεί ροέ χρήματος και πρέπει να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες ε, πέρα από τις εθνικές ε, αρχές ε, και μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών θα μπορούσατε να δημιουργήσετε μια τέτοια σχετική μονάδα στη Europol που αυτομάτως έχει τις πληροφορίες. Απορρίφθηκε στην διαδικασία του τριμερούς διαλόγου και δεν θα μπει στην τελευταία ε, οδηγία, μια απλή πρόταση που νομίζω θα έκανε τη διαφορά. Ευχαριστώ την ε, κυρία Γκραπίνη. Όσον αφορά το θέμα της ασφαλείας, προσπαθούμε ναι. πραγματί να εντάξουμε την κοινότητα και από αυτήν την έννοια θα έπρεπε να αναφέρω την σημαντική διάσταση των διαπραγματεύσεων του Brexit και εγώ δεν θα ήθελα να σχολιάσω. Γεγονός είναι ότι το κράτος μέλος αυτό, όπως και άλλα, παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο να διασφαλίσει την συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης ε, και νομίζω ότι αυτό αναγνωρίζεται κάπως ε, στην λύση που έχουμε. Πάρα πολύ απλά το συλλογικό συμφέρον ασφαλείας ε, της Ευρώπης σήμερα και η φύση των απειλών είναι πάρα πολύ μεγάλες για να αποτύχουμε πρέπει να επιτύχουμε. Γνωρίζω ότι ο χρόνος πιέζει, δεν θα απαντήσω σε όλα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ζαχαρία για... αυτό το οποίο είπε για την ελευθερία και την ασφάλεια. Πάρα πολύ σωστό. Εγώ θεωρώ ότι το ερμηνεύω ως μια εκπαίδευση σε μια κουλτούρα καινοτομίας Είμαστε μια μεγάλη κοινότητα και νομίζω έχουμε και ένα καθήκον να πρωτοπορούμε στον τομέα των ιδεών, να προωθήσουμε μια διαφορετική αντίληψη σε αυτά τα περίπλοκα ζητήματα. Ε, όσον αφορά την ε, Σλοβακία, κάτι άλλο το οποίο είπε η κυρία Τσενίτσκη, δεν γνωρίζουμε ακόμα αρκετά για την έρευνα. Υποστηρίζουμε την υπόθεση κατόπιν αιτήματο των αρχών της χώρας, όπως κάνουμε και στην Μάλτα και δεν ξέρουμε ακόμα τη φύση της υπόθεσης. Τέλος, κύριε Γκίγιομ μίλησε για το πώς μοιραζόμαστε τα δεδομένα. Αναπτύσσουμε τις δυνατότητές μας και την σήμερα ημέρα με την σώματεμπορία και την εκμετάλλευση των γυναικών είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις σας. Για άλλη μια φορά, να σας εκφράσω τη χαρά που είχαμε ως Επιτροπή για τη συνεργασία που είχαμε μαζί σας τα τελευταία 9 χρόνια. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά πάρα πολύ. Yes, Now have prepare voting. Λοιπόν, να προετοιμαστούμε τώρα για την ε, ψηφοφορία. Uh, Συνάδελφοι, ετοιμάστε τις κάρτες της ψηφοφορίας σας παρακαλώ. Να κάνουμε μια δοκιμή, να δούμε ότι τα μηχανήματα μας λειτουργούν. Ψηφίστε παρακαλώ δοκιμαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ε, έλεγχο κάνουμε, έλεγχο. Μια δοκιμαστική λειτουργία να δούμε ότι όλα λειτουργούν σωστά. Ναι, <laughs> okay, thank you Ωραία, σας ευχαριστώ. Και περνάμε στη γνωμοδότηση του κυρίου Άλμπρεχτ για τον κανονισμό για τον ΕΝΙΣΑ, τον οργανισμό για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την κατάρριξη του κανονισμού 526 του 2013, καθώς και για την πιστοποίηση ασφαλείας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφορίας και των επικοινωνιών. Πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Έχουμε πολλούς ε, συμβασμούς. Περνάμε στην πληροφορία. Ε, συμβαστική τροπολογία 1. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 62 δύο. Άρχεται η ψηφοφορία. Close the vote. Πέρας. Κάρετ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 63. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 68. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 69, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 71. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 72. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 78. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Rejected. Απορρίφθηκε. 79. Άρχεται η ψηφοφορία. Close the vote. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 80. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας τη ψηφοφορία. εγκρίνεται. 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 13. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία, τροπολογίες 83 και 84 που ταυτίζονται. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 85. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. sorry. Amendment 15. Τροπολογία 15. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 15. Close the vote. ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται. 92 και 16 που ταυτίζονται. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. εγκρίνονται. 94. Ψηφίστε παρακαλώ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 95. Άρχεται η ψηφοφορία. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 96. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 98. Συμφίστε παρακαλώ. Πέρασε της εγκρίνεται. Όχι, συγγνώμη, απορρίφθηκε. Απορρίπτεται. Yes, I vote with S&D. Probably. That's good. <laughs> I have to change my vote. Mm. Uh, amendment 99. Uh, Τροπολογία 99. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 105. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Rejected. Απορρίπτεται. 106 και 18 από κοινού. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Rejected. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται. Τροπολογία 18. Ψηφίστε. Πέρας φορείες. Εγκρίνεται. 107. Ψηφίστε παρακαλώ, πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 116. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 117. Άρχεται... 17. Άρχισε η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 125. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 10. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 29. Ψηφίζουμε. Ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται. 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 34. Ψηφίστε παρακαλώ για την 34. Πέρας. Απορρίπτεται. 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 37. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 38. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. εγκρίνεται. 39. Ψηφίστε παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 40. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται. 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 43. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 44. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 45. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 46. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Ψηφίστε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 50. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 53. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 54. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα για την 54. Πέρας της Εγκρίνεται. 55. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 58. Όχι, όχι, συγγνώμη. 59. 59. Ψηφίζουμε επί τις τροπολογίες 59. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 60. Ψηφίζουμε. Για την τροπολογία 60. Μέχρι τώρα. Απορρίπτεται. Λοιπόν, ψηφορία επί του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Σας ευχαριστώ. Sorry, I want to change my vote. Uh, εγώ θέλω να αλλάξω την ε, ψήφο μου για την υπαριθμό 94, την ε, τροπολογία, γιατί τελικά μου είχαν σημειώσει εδώ πέρα συν και όχι πλήν. Ευχαριστώ. Okay, dear Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο τμήμα της ε, συνεδρίασής μας. Ε, περνάμε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ε, Τεχνολογίας Πληροφορικής στον χώρο Ελευθερίας, Ασφαλείας και Δικαιοσύνης. Η κυρία η κυρία Μόνικα Μακοβέ είναι η συγγήτρια. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσουμε την εισηγητρία για το πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις ε, για το θέμα αυτό που τον Ιανουάριο πήγε στον ε, τριμερή διάλογο. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαστε στον ε, τριμερή διάλογο, ελπίζουμε να τελειώσει. Έχουμε λοιπόν το τα που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας, το πώς εφαρμόζει την διαλειτουργικότητα, ζητήματα που αφορούν ε, ακριβώς ε, τα τεχνικά σημεία, το τι θα αναθεθεί σε εξωτερικούς εργολάβους και την εφαρμογή τεχνικών λύσεων για να λειτουργούν τα συστήματα 24 ώρες ε, το 24ωρο και 7 μέρες τη βδομάδα. Υπάρχουν λοιπόν πολλές ε, τεχνικές ε, λύσεις και τα συζητάμε ακόμα τα ζητήματα. Αυτό αφορούσε ακριβώς την λειτουργία της υπηρεσίας. Κατόπιν έχουμε τα θέματα διαχείρισης Τη υπηρεσία, ε, δηλαδή τον εκτελεστικό διευθυντή, ε, αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή, σύνθεση διοικητικού συμβουλίου, διαχείριση των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας. Μέχρι στιγμής οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων είναι πολύ επικοδομητικές. Καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία επί πολλών διατάξεων. Ε, κάποια ζητήματα παραμένουν ακόμα υποσυζήτηση, αλλά θεωρώ ότι η οι συγκητές και οι συνομοθέτες θα καταλήξουν σε μια συμφωνία και ελπίζω η επόμενη συνεδρίαση του τριμερούς διαλόγου θα λάβει χώρα τέλη Μαρτίου και να είναι η τελευταία. Ευχαριστώ και την κυρία Κινίτσι που είναι πάντα στην διάθεσή μας και ε, επειδή μας βοήθησε πολύ για να επιτύχουμε συμφωνία. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ Μόνικα ως σκιώδης εισηγητρία να σε ευχαριστήσω και εγώ για τον πολύ ανοιχτό διάλογο. Ναι, ναι, μα εσείς ήσασταν οι μόνοι που ήρθατε. Πάντα, πάντα. Κυρία Τσενίτσα, θέλετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Μόνικα και για τα καλά της λόγια αλλά και για τη δουλειά της. Ήδη μας έχει ενημερώσει για το τι έχει γίνει. Ακόμα υπάρχουν κάποια θέματα πολιτικά που εκκρεμούν, αλλά θα τα λύσουμε στις τεχνικές συναντήσεις. Θα εξευρεθεί πολιτική λύση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό ο κανονισμό γιατί είναι πολύ σημαντικέ και αυτέ οι αρμοδιότητε που αφορούν την ενίσα. Σε ευχαριστούμε και πάλι Μόνικα. Ε, εμείς ευχαριστούμε λέει η πρόεδρος. Και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη των τριμερών διαπραγματεύσεων και τώρα έχουμε τη μελέτη ε, του θεματικού τμήματο δικαιωμάτων πολιτών και υποθέσεων όσον αφορά πολιτικέ και νόμιμε ευρωπαϊκή ένωση και των κρατών μελών για πρόσωπα ύποπτα για εγκλήματα που έχουν σχέση με την τρομοκρατία. Η τύση τη Επιτροπή μα έγινε αυτή η μελέτη και αναλύει το πώ σε 10 κράτη-μέλη δίνεται ορισμό αυτών των ε, ε, υπόπτων και ανταλλάσσουν πληροφορίε και τι μέτρα μπορεί να ληφθούν, ώστε οι αρχέ να, να προβάλλουν και να ερευνήσουν τα σχετικά εγκλήματα. Το κείμενο το έχετε λάβει με την έγγραφα της συνεδρίασης και υπάρχουν και σε χαρτί κάποια αντίτυπα εδώ στην αίθουσα. Και τώρα δώσουμε το λόγο στον κύριο Κόντεν Λίγκερ. Λίγκερ, Λάγκερ. Α, Λιζέ, Λιζέ, Λιζέ. Από την Optimity Advisors και θα σας παρουσιάσω τα βασικά σημεία της έκθεσης. Um, uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε το τμήμα δικαιωμάτων των πολιτών ε, μας ανέθεσε να κάνουμε μια μελέτη για τους νόμους για τα άτομα που είναι ύποπτα τρομοκρατίας. Είχαμε λοιπόν τον Δ. Κάρολιν Μίλλερ, τον Μαξ Χένρι, τον Δ. Γένιο Ζώσμερ Μέρια Γκρούτχαιλ και επίσης είχαμε την βοήθεια κάποιων εξωτερικών συμβούλων. Υπάρχουν κάποια αντίγραφα της έκθεσης ε, δίπλα στην αίθουσα. Η εταιρεία μας ε, κάνει πολλά πράγματα για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ανοίξαμε γραφείο στο Βερολίνο, πριν είχαμε έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Οπότε σήμερα Έχουμε πόσο, 10-15 λεπτά. Α, δεν φαίνονται οι διαφάνειες, δεν πειράζει, εντάξει. Waiting for slides. The slides are very succinct, so we can do without them as well. Κοιτάξτε, είναι λιτά και περιεκτικά, οπότε μπορούμε και χωρίς αυτά. So it's, uh, it's the ε, την επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Λοιπόν, σήμερα θα θέλαμε να καλύψουμε τους στόχους της μελέτης, να δούμε τις τάσεις των τρομοκρατικών επιθέσεων, το νομικό πλαίσιο και μετά να περάσουμε στα πιο ουσιαστικά θέματα, τα δικαιώματα των υπόπτων τρομοκρατίας, ε, μηχανισμούς διαμοιρασμού ε, πληροφοριών ε, εντός και εκτός κρατομέλων και συμπεράσματα. Όπως είπα, η έκθεση είναι διαθέσιμη, 200 σελίδες. Ε, η κυρίως έκθεση είναι 50 σελίδες, τα άλλα είναι παραρτήματα, οπότε θα προσπαθήσω να τα συνοψίσω. Λοιπόν, η ε, στόχη ήταν να δούμε τις σχετικές νομικές διατάξεις που ισχύουν για υπόπτους τρομοκρατίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια γενική εικόνα των υφιστάμενων μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών εντός και εκτός κρατών και να διατυπώσουμε συστάσεις επί τη βάση των ευρημάτων αυτών. Η έρευνα για την έκθεση αυτή έγινε πέρσι δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2017, οπότε κάποια πράγματα έχουν αλλάξει. Εστιάσαμε σε 10 κράτη-μέλη, Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία, Βρετανία, Σουηδία, Ελλάδα, Γερμανία, Ολλανδία. Για κάθε μία από αυτές τις χώρες έχουμε μια ξεχωριστή έκθεση στα παραρτήματα. Και ε, όσον αφορά την μεθοδολογία εστιάσαμε ε, σε συνεντεύξεις ε, στα κράτη-μέλη αυτά, συνεντεύξεις στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ερευναγραφείου και κάποιους ειδικού, όπως είπα. Όσον αφορά δε, τις τάσεις στην τρομοκρατία, τα τελευταία 15-20 χρόνια είχαμε κάποια αλλαγή στις ε, τάσεις. Α, το ξέρετε βεβαίως είναι δύσκολο να μιλήσουμε για στατιστικά στοιχεία τρομοκρατίας ε, λόγω διαθέσιμότητας των δεδομένων, αλλά υπάρχει μείωση από τη δεκαετία του 70 και 80 στον αριθμό τρομοκρατικών ε, χτυπημάτων, αν και τα τελευταία χρόνια είχαμε μία αύξηση. Επίσης υπάρχει μια αλλαγή στην φύση της ε, τρομοκρατίας. Έχουμε φύγει από το χαρακτηριστικό της ε, δεκαετίας 70, 80 και 90 εθνικιστικών κινημάτων, ΕΤΑ, IRA και αναρχοαριστερής τρομοκρατίας, με φραξιών, οι αριθρές ταξιαρχίες ε, και τα ανάλογα στο Βέλγιο και τα τελευταία χρόνια έχουμε τζιχαντιστική τρομοκρατία και δεξιά τρομοκρατία, υπόθεση Breivik, αλλά και ο απερχόμενος αρχηγός της Ρετρομοκρατίας του Ηνωμένου Βασίλειο είπε ότι το 2017 ε, είχε αποτρέψει τέσσερις τέτοιες επιθέσεις ε, το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες αλλάζουν. Υπάρχει μια αύξηση στον αριθμό βομβών ε, και κρίξεων. Επίσης οι δολοφονίες ε, αποτελούσαν το 27% των ε, επιθέσεων ε, τη δεκαετία του 70, τώρα είναι 1% το 16 και 17 και είχαμε αύξηση των ένοπλων επιθέσεων από 7% στη δεκαετία του 80 και πήγαν στο 15% μεταξύ 2010-2016. Επόμενη διαφάνεια. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες ε, σε ζητήματα τρομοκρατίας, νομίζω ε, τα ξέρετε μάλλον καλύτερα από μένα, περιορισμένες ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς υπάρχει το άρθρο 3 παράγραφος 2 τη συνθήκη της Ένωσης που λέει ότι η Ένωση θα παρέχει μια περιοχή ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και το άρθρο 83.1 τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που αναφέρει διάφορα αδικήματα για τα οποία μπορεί να επιβάλλει κάποιο ελάχιστο κανόνε η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των οποίων τρομοκρατία. Ε, όσον αφορά την κοινή νομοθεσία υπάρχει η οδηγία για την καταπολέμηση τη Τρομοκρατία που πέρασε πέρσι νομίζω και τα κράτη-μέλη πρέπει να τη μεταφέρουν μέχρι το Σεπτέμβριο. Προφανώς ε, είναι το βασικό μέσο, έχει έναν ορισμό της δημοκρατίας που είναι αρκετά ενδιαφέρον και όσον αφορά λοιπόν τη δευτερογενή νομοθεσία υπάρχει ένας αριθμός μέσων που εστιάζουν όχι αποκλειστικά στη δημοκρατία, αφορούν αυτά τα οποία ανέφερα, την ε, οδηγία καταπολέμησης ε, του ξεπλήματος χρήματος, διαλειτουργικότητα και μεγάλα ε, συστήματα πληροφορική και αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα έγγραφα μετά, όπως η στρατηγική, η στρατηγική του 2005 για την τρομοκρατία και η Ευρωπαϊκή Ατζέντα του 15 για την ασφάλεια. Αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι η εθνική ασφάλεια παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, όπως αναφέρει το άρθρο 4 παραγωγής 2 της συνθήκης. Και θα επανέλθουμε σε αυτό όταν μιλήσουμε για την ανταλλαγή πληροφοριών. Μιλάμε για ένα φαινόμενο διασυνοριακό που οι αρμοδιότητες ε, παραμένουν στο εθνικό επίπεδο. Να δούμε λοιπόν την επόμενη διαφάνεια τα δικαιώματα των υπόπτων τρομοκρατίας. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια ποινικοποίηση των σχετικών αδικημάτων, η οποία έχει διευρυνθεί. Παραδείγματο χάρη ε, έχουμε προχωρήσει πέρα από την ίδια την τρομοκρατική δράση, δηλαδή κάποια πρόδρομα αδικήματα παρότρινση σε τρομοκρατία, ταξίδι με σκοπό την εκπαίδευση, την τρομοκρατική ή στοιχεία προετοιμασίας ε, τρομοκρατικής δράσης, τα οποία ε, ποινικοποιούνται και αυτά. Ταυτόχρονα υπάρχει μια αύξηση των ε, διοικητικών αρμοδιοτήτων για πρόληψη και ποινικοποίηση τέτοιων συμπεριφορών. Αυτή είναι μια τάση που υπάρχει νομίζω σε όλες τις χώρες που βλέπουμε. Με παραδοσιακή νομίζω έτσι, εποπτεία, ε, δικαστική εποπτεία. Η Σουηδία έχει αρκετά ισχυρή δικαστική εποπτεία. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα όμως, κάποια από τα στοιχεία όπως η αφαίρεση ταξιδιωτικών εγγράφων ε, για να μην μπορεί ένας ε, τρομοκράτης ή μάλλον Επίδοξο τρομοκράτη να ταξιδέψει. Αυτό είναι διοικητικό και όχι δικαστικό μέτρο. Ω παράδειγμα, περιορισμό ε, της ελευθερίας ε, μετακίνησης ε, σε κάποια κράτη-μέλη. Ο νόμος λέει ότι περί κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στην Γαλλία προβλέπει ότι μπορεί να περιοριστούν στα όρια ενό Δήμου, παραδείγματο χάρη. Και να σα δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Στην Ολλανδία ένα άτομο απαλλάχθηκε από δικαστήριο από την κατηγορία τρομοκρατικών δραστηριοτήτων λόγω έλλειψης αποδεκτικών στοιχείων. Και όμως μετά την αθώση του, του επιβλήθηκαν διοικητικά μέτρα για να μην ταξιδέψει σε κάποιες περιοχές του Ρότερνταμ κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου ένα παράδειγμα διοικητικών μέτρων που ε, εξαπλώνονται. Επόμενη διαφάνεια, αυτό το οποίο παρατηρήσαμε και βρήκαμε είναι μια κατάταξη ε, διαφόρων δικαιωμάτων ε, ανάλογα με τα άτομα. Έχουμε τα δικαιώματα που έχει ο κάθε ύποπτος ή κατηγορούμενος όταν έχει ξεκινήσει η ποινική διαδικασία. Αυτό είναι το εύκολο δηλαδή όλοι όσοι εμπλέκονται σε μια τέτοια διαδικασία. Έχει κάποια δικαιώματα, κάποια είναι στο πακέτο δικαιωμάτων υπόπτων. Υπάρχουν ίσως ε, κάποια ζητήματα που αφορούν ιδιαίτερα την τρομοκρατία. Παραδείγματο χάρη έχουμε το καστός απομόνωσης ε, στην Ισπανία. Στην Γαλλία η προφυλάκηση μπορεί να επεκταθεί μέχρι και σε τέσσερα χρόνια σε περίπτωση τρομοκρατίας ενώ συνήθως είναι τρία χρόνια. Μετά υπάρχουν τα δικαιώματα των ατόμων τα οποία υφίστανται διοικητικά μέτρα, όπως σας είπα. Ανάκληση διαβατηρίου και συχνά ενώ υπάρχει βεβαίως ε, η δυνατότητα δικαστικής προσφυγής, η δικαστική εποπτεία της διαδικασίας που οδηγεί στα διοικητικά μέτρα ε, είναι ad hoc, δηλαδή μπορεί να γίνει μόνο αφού επιβληθούν τα διοικητικά μέτρα. Αλλά και πάλι ο ύποπτος γνωρίζει ότι ε, υφίσταται τέτοια μέτρα. Μετά περνάμε σε κάτι το οποίο είναι μάλλον γκρίζα ζώνη και αφορά τα άτομα ενδιαφέροντος, ας τα πούμε, άτομα τα οποία παρακολουθούνται είναι στο ραντάρ ας πούμε των αρχών και μπορεί να μην το γνωρίζουν, μπορεί να παρακολουθούνται τα τηλεφωνήματά τους στη Γαλλία παραδείγματος χάρη ναι. θα ήταν ε, κάποιος ο οποίος έχει φάκελο S ε, στην ασφάλεια δηλαδή και το πρόβλημα με αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι τα άτομα δεν γνωρίζουν ότι αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος των αρχών μέχρι να υποστούν κάποια διοικητικά μέτρα ή ποινικέ διαδικασίες. Και τέλος, έχουμε τα δικαιώματα που έχει οποιοδήποτε βρίσκεται στην επικράτεια της Ένωσης και αρκετέ από τις μεθόδους που ανέφερα ε, αφορούν οποιονδήποτε από εμά αντί για ε, άτομα με τα οποία είναι ύποπτα τρομοκρατίας ε, π.χ. η δυνατότητα εξακρίβωσης των στοιχείων στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει επεκταθεί τώρα και η αστυνομία μπορεί να σταματήσει τον οποιονδήποτε χωρί να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη υποψία. Το, η κατάσταση εκτάκτου ανάγκη στην Γαλλία επίσης επιτρέπει πιο παρεμβατικές μεθόδους όσον αφορά τον περιορισμό της κίνησης εντός της επικράτειας. Παρακατώ τώρα. Η άλλη διαφάνεια. Εν μετρό της ε, πληροφορίες των κρατών μελών, κάτι το οποίο σχετίζεται με αυτές τις τέσσερις κατηγορίες που αναφέραμε γιατί πρόκειται για κάποια μέτρα τα οποία είναι δοκιμασμένα για την ανταλλαγή πληροφόρηση σε κάποιες ε, περιπτώσεις όσον αφορά κάποιες έρευνες που διαρκούν και τώρα έχουμε αυτή τη φιά ζώνη μεταξύ δράση διοικητικών αρχών και υπηρεσιών πληροφοριών. Και αυτό σε διεθνές επίπεδο αφορά και τις τρίτες χώρες. Νομίζω σας τα είπε ο κ. Γουίνραντ προηγουμένως ότι έχουμε Ε, κάποιες ξεκάθαρες μεθόδους ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά από την έρευνα πρόκειψε στο ότι οι αρχές στηρίζονται και σε άτυπες μορφές ανταλλαγής πληροφοριών και αυτό διεθνώς. Το οποίο βέβαια έχει κάποιες επιπτώσεις στο πρωτοδικαστικό έλεγχο και αυτό έχει σχέση και με το να γίνει γνωστό το αν κάποιο ε, είναι όντω ύποπτο και τι δραστηριότητες έχει αναπτύξει. Α, για να δούμε τώρα καταληκτικά. Έχουμε βέβαια και άλλα συμπεράσματα και άλλες συστάσεις στο κείμενο. Πάντως το πρώτο θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ε, συμφωνία για το ποιο είναι ο ορισμός του υπόπτου και αυτό έχει συνέπειε σε σχέση με το αρχικό ερώτημα δηλαδή για το ότι δικαιώματα έχουν οι ύποπτοι για τρομοκρατία και συναφή εγκλήματα. Ε, επίσης τα κράτη-μέλη τείνουν να αντιμετωπίζουν τους υπόπτους εκτός ποινικής δικονομίας με διοικητικά μέτρα και κυρώσεις. Ε, αρκετοί είπαν <coughs> ότι τώρα είναι ο κανόνας ε, η η έκτακτη αντιμετώπιση και τον Νοέμβριο του 2017 είχαμε νέο νόμο στην Γαλλία ούτω ώστε να παραταθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που είχε επιβληθεί μετά την επίθεση στον Πατακλάν. Βέβαια, το θέμα είναι πόσο αποτελεσματικά είναι αυτά τα μέτρα τι γίνεται με την ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα και σα παραμείνουμε στον Οφλάχερντε, στον επικεφαλής της Υπηρεσία τα ανθρώπινα δικαιώματα που συχνά λέει ότι τα βασικά δικαιώματα βρίσκονται στην καρδιά οποιοδήποτε δήματο και θα πρέπει εκ των υστέρων να τα σκεπτόμαστε ακόμα και για θέματα ασφάλεια. Εν προκειμένου λέμε ότι θα πρέπει να δούμε τα δικαιώματα των υπόπτων. Πολύ σημαντικό και σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς λέει η πρόεδρος. Και τώρα συζήτηση. Ποιος θέλει το λόγο. Κυρία Σίπελ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και για τη μελέτη. Πάντως έχω προβληματιστεί γιατί ήλπιζα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για να μας βοηθήσετε στη δουλειά μας στο τέλος της παρουσίασης μας είπατε για τους υπόπτους. Επί ποιες βάσεως χαρακτηρίζεται κάποιος ύποπτος και πιθανά τρομοκράτες εάν δεν υπάρχει κοινή βάση, κοινός ορισμός. Όμως Υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών για κάποιον που θα μπορούσε να είναι τρομοκράτη. Ε, τότε δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση αυτή. Πώ υπάρχει έτσι αμοιβαία εμπιστοσύνη, πώ υπάρχουν αρκετέ πληροφορίε προ τούτο. Βέβαια υπάρχει υποψία, αλλά δεν υπάρχουν ε, απτά αποδεικτικά στοιχεία. Γιατί αν υπάρχουν τότε πάμε στην ποινική αντιμετώπιση. Αλλά σύμφωνα με τη μελέτη σα αυτό όλο ένα και περισσότερο δεν συμβαίνει. επομένω ας πούμε ότι εκρεμεί κάποια υποψία. υποψία εναντίον σας μπορεί να μην ε, είναι αληθής, αλλά πώς θα αποδείξετε ότι είναι αναληθής αυτή η κατηγορία. Πόσο καιρό θα σας παρακολουθούν, πόσο καιρό θα έχετε περιορισμό στην ελευθερία διακίνησή σας, μα πώς θα αποδείξω ότι δεν είμαι ή δεν είσαστε ένοχος και ότι δεν κάνατε τίποτα. Οπότε αυτό παραπέμπει στο γενικότερο πρόβλημα δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Επίσης και κάτι άλλο με προβληματίζει. Κάποια μέτρα που λάμβανε σε κάποια κράτη μέλη, που όταν μας μιλήσατε για αυτά τα τέσσερα χρόνια που χρειάζεται κάποιος για να προσβιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου. Δηλαδή, χρειάζεται τόσο πολύ κάποιος να, έχει, να είναι σε, σε, σε είδους προφυλάκηση και να πάει μετά στο δικαστήριο ή να μην πάει ποτέ. Ε, πολύ σημαντικό και αυτό. Δεν ξέρω, μπορείτε να επισέλθετε σε λεπτομέρειες. Για ποινικοποίηση κάποιων συμπεριφορών. Ποιων συμπεριφορών. Είπατε για τον περιορισμό του δικαιωματικού διακίνηση, του. Ε, αναστολή, αφαίρεση τέλο πάντων διαβατηρίου και άλλες ε, κυρώσει. Μα υπάρχει σαφής διάκριση ούτω ώστε να ξέρουμε ποια συμπεριφορά επισύρει τέτοιες κυρώσει. Α, και το τελευταίο για τη μελέτη σας. Ποιοι ήταν οι εμπειρογνώμονες από τους οποίους ενημερωθήκατε δικαστικές αρχές, αστυνομικές αρχές, νομικούς, ειδικού για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι, τι, ποιοι ήταν. Ε? Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να έχει ζητήσει κάποιο άλλο το λόγο, οπότε δίνω το λόγο στον προσκεκλημένο να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα αλλά σας καλώ να διαβάσετε και την μελέτη. Να ξεκινήσω με το τελευταίο ερώτημα. Έχουμε έναν κατάλογο με τους ανθρώπους ή με, το, με τις ιδιότητές τους ε, που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις. Σε αυτές τις μελέτες συνήθως είναι πιο εύκολο να κάνεις συνεντεύξεις με ανθρώπους από την, από την δικαιοσύνη, ή ε, ε, νομικούς, γιατί πιο, πιο δύσκολο είναι να έχεις πρόσβαση στους ανθρώπους που δουλεύουν στις αρχές επιβολής του νόμου. Οπότε ε, σίγουρα ε, πιο πολλές προφορές αντλήσαμε από τη δικαστική εξουσία. Αν και προσπαθήσαμε να αντλήσουμε όσο την δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και από πανεπιστημιακούς, από εμπειρογνώμονες. Συγγνώμη τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το, το όνομα. για παράδειγμα τον Σον Μέρφυ με τον οποίο μιλήσαμε, πανεπιστημιακό, γιατί ακριβώς οι πανεπιστημιακοί μπορούν να μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα για την πλευρά της επιβολής του νόμου. Οπότε παίρνουμε υπόψη μας όλες αυτές τις διαστάσεις όταν εκπονούμε αυτές τις μελέτες. Για να είμαι ειλικρινής, τα, άλλα ερωτήματά σας είναι πολύ δύσκολα να τα απαντήσω. Γιατί, όπως γνωρίζετε, η νομοθεσία ε, για τις, ε, για τις τρομοκρατικές πράξεις συνήθως ε, καθοδηγείται κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις. Δηλαδή υπάρχει ένα τρομοκρατικό περιστατικό και στη συνέχεια λαμβάνονται νομοθετικά μέτρα. Αυτό συνδέεται πολλές φορές και με έναν ιδιαίτερο συναστηματισμό ακριβώς γιατί προσπαθεί η νομοθεσία να απαντήσει στις ανησυχίες της κοινή γνώμης δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια και όχι τόσο στα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Γαλλία και η κατάσταση εκτακτής ανάγκη που έχει επιβληθεί εκεί είναι πλήρω αποδεκτή πλέον στην κοινή γνώμη ε, και ο νόμος που πέρασε στα τέλη της περσής χρονιάς δεν θα είχε περάσει ποτέ πριν από κάποια χρόνια αλλά ακριβώ επειδή έγιναν όσα έγισαν στην ε, Γαλλία η κοινή γνώμη έχει αλλάξει στάση, έχει υπάρξει μια μεταστροφή. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του υπερασπιστή των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ακριβώς ε, λόγω αυτής της, ε, αυτής της αμφίροπης ισορροπίας που υπάρχει ανάμεσα στην ασφάλεια και τις ελευθερίες. Γιατί πολλοί, πολλοί πολίτες ενδιαφέρονται πιο πολύ για την ασφάλειά τους αυτή την περίοδο. Για το βάρος της απόδειξης και για το πώς μπορεί κανείς να αιτιολογήσει ή να απαντήσει στο γιατί δεν είναι ένοχο ή δεν θα έπρεπε να είναι ύποπτο τρομοκρατία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το ερώτημα. Ένα, θέμα το οποίο ήθελα να θέσω, το είχα στη διαφάνεια, είναι ε, η ανάγκη να υπάρχουν περισσότερε πληροφορίε, περισσότερα δεδομένα. Γιατί ε, αυτό που κάνουμε ε, σε τέτοιε μελέτες είναι να κοιτάμε αριθμού Στη Γαλλία αναφέρομαι συχνά στη Γαλλία γιατί την ξέρω πολύ καλά την περίπτωση αυτή. 6.000 έρευνε έγιναν έπειτα από την επιβολή της έκτακτης, ε, κατάστασης ανάγκη. ανάγκης. 21 συλλήψει έγιναν και αυτό από τη στιγμή, από την επιβολή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης ε, από 1η Νοεμβρίου, δηλαδή πέρσι. Νομίζω ότι ο διαμερισμό στοιχείων ε, όσον αφορά τις τρομοκρατικέ επιθέσει ή τα θύματα τη τρομοκρατία, θα μας βοηθούσε για να σχηματίσουμε μια καλύτερη εικόνα της αναλογικότητας της απάντησης που δίνεται, διότι προφανώς υπάρχει ανάγκη να εξασφαλίζεται η ασφάλεια, αλλά υπάρχει και μια διάσταση θεμελιωδών δικαιωμάτων που κάποιες φορές την ξεχνούν οι αρχές και είναι πολύ εύκολο να την ξεχνούν. Και ε, δυστυχώς το πρόβλημα είναι ότι άπαξ και ξεχάσει κανείς τη διάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι πολύ δύσκολο να την επαναφέρει κανείς. Αυτά ήταν δύσκολα τα ερωτήματά σας, αλλά είμαι στη διάθεσή να συζητήσουμε περαιτέρω αν θέλετε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σαρτζεντή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις να θέσω. Πρώτον, υπάρχει ένας ευρύτερος ορισμός που έχει προταθεί στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και αφορά την τρομοκρατία. Εσείς από τη μελέτη σας διαπιστώσατε ότι υπάρχουν ύποπτοι οι οποίοι είναι ύποπτοι λόγω της ευρύτερης, του ευρύτερου αυτού ορισμού της τρομοκρατίας που παλαιότερα δεν θα ήταν ύποπτοι τρομοκρατίας. Για παράδειγμα, άνθρωποι που προκαλούν οικονομική ζημία σε ένα κράτος ή περιβαλλοντικοί ακτιβιστές, τέτοιου είδους κατηγορίες ανθρώπων εννοώ. Αν έχετε διαπιστώσει κάτι τέτοιο, το ερώτημά μου, και το άλλο ερώτημα είναι όταν ένας αστυνομικός ε, κάνει έλεγχο στο δρόμο, ε, ίσως ε, σε αναγκάσει να ανοίξει το πορπαγκά σου για παράδειγμα, ενώ οδηγεί το αυτοκίνητό σου. Από πότε ένας απλός έλεγχος, μια διαπίστωση στοιχείων γίνεται έρευνα, διότι όταν υπόκεισε σε έρευνα, σε ανάκριση, τότε έχεις δικαίωμα να απευθυνθείς και σε δικηγόρο. Και ε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση να υπάρχει, όπως είπατε και εσείς, ε, να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι και αντίστοιχα να αυξάνονται και οι περιπτώσεις ε, προανάκρισης. Υπάρχει δηλαδή μια ευθεία σχέση. Μήπως μπορείτε να μας πείτε περισσότερα στοιχεία γι' αυτό. Για τον ευρύτερο ορισμό της τρομοκρατίας, όπως είπα, Νομίζω ότι η οδηγία για την τρομοκρατία θα πρέπει να, μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι το τέλος του 2018. Έχουμε, δεν έχουμε δει δηλαδή ακόμα συγκεκριμένα στοιχεία. Ένα γαλλικό παράδειγμα να σας ξαναδώσω. Είναι η διάσκεψη για το, για το κλίμα που έγινε στο Παρίσι, 21, που έγινε λίγες μέρες μετά την επιβολή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Γαλλία. Και υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι οι αστυνομικές αρχές ε, αξιοποίησαν τις ε, αρμοδιότητες που τους δόθηκαν προκειμένου να περιορίσουν την κίνηση, την κυκλοφορία ακτιβιστών ε, που δεν είχαν σκοπό βεβαίως να διαπράξουν τρομοκρατικές ενέργειες και ακριβώς χρησιμοποιήθηκαν αντιτρομοκρατικοί νόμοι. Επίσης υπάρχουν τομείς όπου η γαλλική ε, αστυνομία μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει αντικρομοκρατική νομοθεσία στη Δουνκέρκη. Εγώ δεν είμαι ε, ειδικό ε, σε ζητήματα τρομοκρατίας βεβαίω, αλλά νομίζω ότι το λιμάνι της Δουνκέρκης δεν είναι και το, το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη πύλη εισόδου ε, τρομοκρατών, αντίθετα άλλα ζητήματα ε, χαρακτηρίζουν το λιμάνι αυτό. Τι, τι ακριβώς έγινε, ρωτάει η κυρία Σαρτζεντίνη, στη Δουνκέρκη. Εκεί η αστυνομία χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση τις εξουσίες που, τους έχει, που τις έχει χορηγήσει η αντιτρομοκρατική νομοθεσία. Τώρα, αν πράγματι υπάρχει ένα σκεπτικό για το γιατί γίνεται αυτό στη Δουνκέρκη και ενδεχομένω αλλού ή όχι ε, είναι, είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Ε, ε, η κυρία Σατζεντή ρωτάει, σχετίζεται με τη μετανάστευση προφανώς από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Πιθανότατα, απαντά ο μιλητής. για το άλλο σας ερώτημα. Είναι δύσκολο να το απαντήσω. Ακριβώς διότι αντιμετωπίσαμε δυσκολίες στο να μιλήσουμε με αρχές επιβολής του νόμου, ιδίως αυτές που δραστηριοποιούνται επί τόπου. Αλλά δεδομένου αυτού, αυτή η ρευστότητα ανάμεσα στο, ε, στο να, να σου ψάξουν το αυτοκίνητο να σου ζητήσουν την ταυτότητα και να περάσει στη φάση της ανάκρισης, πράγματι είναι πάρα πολύ θολά τα όρια μεταξύ αυτών των δύο καταστάσεων. Ε, δεν, δυστυχώς δεν, επικεντρωθήκαμε πολύ στην ε, μελέτη μας. Ε, είναι όμως πράγματι μια από αυτές τις γκρίζες περιοχές όπου καλό είναι να, ε, να μελετηθούν, που καλό είναι να μελετηθούν περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να ζητά κάποιος άλλος το λόγο. Επομένως θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Με ενημέρωσαν ότι έρχεται και ο συγητής μας για το επόμενο θέμα. Ε, θα κάνουμε ένα μικρό πεντάλεπτο διαλυματάκι και σε πέντε λεπτά συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λιζέρ για την εξαιρετική παρουσίασή σας και τις πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις που μας δώσατε. <laughs> Uh, dear 13 uh, Στις 13 Μαρτίου, συνάδελφοι, οι συντονιστές συνεφώνησαν να γίνει αυτή η έκθεση για την λειτουργία της περιοχής Σέγγεν. Ακόμη υπάρχουν θέματα όσον αφορά τη λειτουργία της ζώνης Σέγγεν. Ακριβώς με την έκθεση θέλουμε να κάνουμε μια καταγραφή του πώς έχει η κατάσταση και τα διάφορα προβλήματα και ελπίζουμε να ακολουθήσουν και άλλες εκθέσεις. Οπότε έτσι να υλοποιηθεί ο ελεγκτικός ρόλος του Κοινοβουλίου στις 20 ε, Φεβρουαρίου έγινε μια ακρόαση σχετικά και σήμερα θα παρουσιαστεί το σχέδιο του κειμένου και γι' αυτό θα δώσουμε το λόγο στον συντάκτη για κατόπιν στους ε, σκιώδες εισηγητές Κάρλος. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σας τα πω στα πορτογαλικά και σύντομα. Σήμερα έχουμε αυτήν την πρώτη έκθεση του Κοινοβουλίου για το Σέγγεν. Σέγγεν σημαίνει ελευθερία διακίνησης και είναι κάτι πολύτιμο για τους Ευρωπαίους, αλλά έχει και ε, οικονομική διάσταση. <clears throat> Γιατί Πρόκειται για κατάρριξη των συνόρων, πρόκειται για 50 δις ευρώ που κερδίζουμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό για οικονομία, για, για απασχόληση. Ε, οι απλουστευτικές απόψεις δεν ωφελούν. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα. Ε, αυτά ε, διαπραγματεύεται αυτή η έκθεση και επανέρχεται τώρα στο θεματολόγιο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων Ξέρουμε τι πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά όχι τι ε, θέλει το Συμβούλιο. Τώρα επίκειται το Συμβούλιο Υπουργών Ιστορικών και είναι πάρα πολύ σημαντικό επί Βουλγαρικής Προεδρίας να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, πώς θα λυθούν αυτά τα προβλήματα, να εξομαλυθεί η κατάσταση και μέσω αυτής της εκθέσης παρουσιάσαμε τις απόψεις μας. Να σας το πω τώρα ή στα αγγλικά τα υπόλοιπα να σας εξηγήσω πώς καταλήξαμε στα της εκθέσεως. Ακριβώς όπως είπατε, κυρία Κοντίτσκε πέρσι, ξεκίνησε με αυτή τη διαδρομή. Πώς θα κάνουμε πιο ευρωπαϊκό το Σέγγεν, εγκρίναμε ένα νέο μηχανισμό λειτουργίας, αναβαθμίσαμε την Επιτροπή και τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου και κατά συνέπεια είπαμε να συγκροτήσουμε μια ομάδα εργασίας. Προεδρεύω εκεί για να δούμε τι έχουμε πετύχει σε διαφορετικούς τομείς. Με αυτή την ε, έκθεση ελπίζουμε ότι θα αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο ρόλο του Κοινοβουλίου που εκπροσωπεί τους πολίτες. Δεν ήταν και πολύ παλιά που θεωρούσαμε ότι πρόκειται για κάτι εγκριτό και απαραβίστο, πρόκειται για κάτι που αποκλειστικά το χειρίζονται τα κράτη-μέλη, όμως είναι κάτι που έχει επιπτώσεις για τη ζωή του κόσμου. Και την τελευταία τριετία υπήρχαν πολλές δυσκολίες, μεγάλη πίεση. Αυτή την ε, τριετία είχαμε περισσότερους ε, ελέγχους των ιστορικών συνόρων από όσο την προηγούμενη δεκαετία. Ε, σε σχέση με αυτό, όπως τα λέω στην έκθεση ξεκάθαρα, ότι είναι υποπίεση το Σέγγεν. Γιατί το κοινό σύστημα ασύλου έχει καταρρεύσει, δεν εφαρμόζεται το κεκτημένο από τα κράτη-μέλη. Και διαπιστώσαν πολλά προβλήματα στην ομάδα εργασία για αυτά. Εξωτερικά σύνορα, αστυνομική συνεργασία, δικαστική συνδρομή, ποινικέ διαδικασίε, ανταλλαγή πληροφοριών, όλα αυτά τα λέμε στην έκθεση. Ακόμα πιο ανησυχητικό το ότι έχουν εγκριθεί διάφορα μέτρα όπως τα νέα συστήματα πληροφοριών, συστηματική έλεγχη επίσης έχουν θεσπιστεί εις βάρος τέλος πάντων επί πολιτών της Ένωσης. Μα υπάρχουν νέες ε, απειλές. Αλλά θα πρέπει τα κρατημέλη να χρησιμοποιήσουν τα προβλεπόμενα εργαλεία και μέσα. Τα λέμε αυτά στην έκθεση και ξεκαθαρίζουμε ότι το Συμβουλίο θα πρέπει να ακολουθήσει τη γνώμη του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να εγκρίνει μια διαπραγματευτική εντολή για τα σχετικά, γιατί είναι απαράδεκτο να έχει μπλοκαριστεί η νέα υπηρεσία, ενώ υπάρχει πολιτική συμφωνία πριν από 9 μήνες. Όλα αυτά αποτελούν πίεση προς το Σέγγεν. Ε, πιο εύκολο είναι κανεί να κατηγορεί την ελεύθερη διακίνηση παρά να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Ήταν λαϊκιστική προσέγγιση και γι' αυτό και θεσπίστηκαν εσωτερικοί έλεγχοι. Οπότε και τα κρατημέλη παίζουν με τη φωτιά κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει συντονισμός. Δεν υπάρχουν στοιχεία για να γίνει μια σωστή αξιολόγηση. Και τώρα επομένω έχουμε και παράκαμψη των κανόνων λειτουργίας. Αυτό είναι παράνομο. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι να κάνει και με μεγάλη προσοχή να προχωρήσει στο θέμα της ρύθμισης αυτών των εσωτερικών ελέγχων και αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις νέες απειλές, τα νέα προβλήματα για την ασφάλεια. Δεν θα πρέπει όλα αυτά να είναι φτιασίδια για την παράταση των εσωτερικών ελέγχων. Νομίζω ότι θα πρέπει να αποτελεί το Σάγγεν ένα εργαλείο υπέρ των πολιτών, να υποστηρίξουν την Επιτροπή προς αυτή την κατεύθυνση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι αυτά φρενάρουν την πρόοδο. Κύριε Πρόεδρε, εν κατακλείδη, θέλω να σου πω άλλα δύο ε, σημεία. Πρώτον, να ευχαριστήσω για τη συνεργασία των κύριων Σάιφαρα και του κύριου Χόλστερ. Και βέβαια, τον Μάικλ, ε, την Κάθλιν, όλους τους ε, συνεργάτες μας και επίσης θέλω να σας τονίσω ότι με αυτή την έκθεση θέλουμε να αντικατοπτρίζονται στο κείμενο όλες οι επαφές της ομάδας για το Σέγγεν. Και ευχαριστώ την ομάδα εργασία για τη συνεργασία τους και θα συνεργαστούμε τους και ηγητές ούτως ώστε να έχουμε μια ευρεία συνένεση πάνω στο θέμα. Πιστεύω ότι θα πρέπει το μήνυμα να είναι ξεκάθαρο σε σχέση με το Σέγγεν. Και ευχαριστώ. Ε, εμείς ευχαριστούμε. Κάρλος, κύριε ε ευχαριστώ πρόεδρε. ευχαριστήσουμε τον Κάρλος Έλιο για τη δουλειά του, αυτή την πρώτη απόπειρα που κάνουμε. Ε, ξέρει το θέμα. Είναι προοδευτικές για απόψεις που διαμορφώθηκαν για το πόσο χρειάζεται να περισωθεί, να συνεχίσει να υπάρχει ο χώρος Σέγγεν. Προς τα εκεί θέλουμε να πάμε. Είμαι η Ασκιώδης εισηγήτρια, θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και εγώ θα ασχοληθώ με τον κώδικα Σέγγεν, το μηχανισμό αξιολόγηση, το σύστημα πληροφορία Σέγγεν. Και θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πολιτικές που σχετίζονται με το Σέγγεν. Τι γίνεται με την αναβάθμιση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, ε, τη στατική ολοκληρωμένου ελέγχου των σύνορων, τι γίνεται με τη ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα, το θέμα της αιτιολόγησης αυτών των ελέγχων όπως είπατε θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπαθίες μας για τα εξωτερικά σύνορα όλα τα θεσμικά όργανα χωρίς να παρεμποδίζει η ελεύθερη διακίνηση στο εσωτερικό της ε, Ένωσης. Εμπιστοσύνη και ελεγγύη κρατών μέλων το τι κάνουν οι την ιστορική ασφαλεία τα κρατη Και επίσης θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να συμφωνήσουμε για μια αλλαγή του συστήματος που έχει σχέση με το άσυλο που θα πρέπει να γίνεται περισσότερη αλληλεγγύη και να περνάει μέσα από το Σέγγεν. πολλές φορές δεν εφαρμόζονται οι κανόνες του Σέγγεν παρά τους στόχους που έχουν δει σε επίπεδο ένωσης. Ε, επίσης, θα πρέπει να συνεργαστούμε με τα τρίτα κράτη για την μετανάστευση. Και θα πρέπει παρά το ότι δεν μας έγινε τεθεριτός, να μας απασχολήσει και αυτό. Αυτά όσον αφορά την πρώτη παρουσίαση του σχεδίου κειμένου. Ε, ευχαριστούμε. Thank Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την εξαιρετική του έκθεση. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε να προτείνουμε στους πολίτες. Να επαναφέρουμε την σημασία του δημοκρατικού ελέγχου της αποκατάστασης του χώρου Σέγγεν και της επαναφοράς του σε πλήρη λειτουργικότητα. Ευχαριστώ λοιπόν για άλλη μια φορά Κάρλο για το εξαιρετικό σου έργο και για τις ηγετικέ σου ικανότητες ε, στην ε, ομάδα εργασίας, στην οποία συμμετέχω βεβαίως, ε, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να προσέλθω σε όλες τις συνεδριάσεις της, παρά μόνο εξ αποστάσεως σε κάποιες. Το να επαναφέρουμε την ε, λειτουργικότητα του χώρου Σέγγεν προς όφελος των πολιτών είναι ανάγκη και αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης οπτικής για τη λειτουργία της Ευρώπης σήμερα. Και η ελεύθερη κυκλοφορία εντός Ευρώπης, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύω ότι πρέπει να εξασφαλιστεί και στο μέλλον. Όμως η εισαγωγή συνοριακών ελέγχων σε κάποιες χώρες και στη δική μου ε, έθεσε υποδοκιμασία των χώρων Σέγγεν. Και δυστυχώς ε, υπό το φως αυτής της κατάστασης δεν μπορούμε να πούμε πολλά ακόμη. Ε, φαίνεται ότι η συνοριακή αυτή έλεγχη πλέον δεν είναι καθόλου προσωρινή. Ε, υπάρχουν κράτη-μέλη που χρησιμοποιούνται του ελέγχους ακόμη και εκεί όπου δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει ανάγκη πλέον. Και θέλω να παραλάβω αυτό που είπε ο Επίτροπος Αβραμόπουλος πριν από λίγες εβδομάδες, ότι η συνοριακή έλεγχη δεν πρέπει να είναι εσωτερικό ζήτημα. Δεν πρέπει να είναι. Και νομίζω ότι ε, ε, δεν πρέπει να θέτουμε σε κίνδυνο το Σέγγεν. Γιατί ακριβώς αυτό κάνουμε. Ε, από την εισρωή μεταναστών ε, έχουμε περάσει στην, ε, στο, στην ασφάλεια ως ζήτημα χωρίς να αιτιολογείται κάτι τέτοιο από την ίδια την πραγματικότητα. Η έκθεση που έχουμε σήμερα μπροστά μας επισημαίνει την ανάγκη τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τους ισχύοντες κανονισμούς και καλεί την Κομισιόν να αναλάβει ταχεία δράση εναντίον των κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν τους κανόνες. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει ο εισηγητής. Είναι απόλυτα αναγκαίο να μην υπάρχει καμία ανοχή σε τετοιου είδους συμπεριφορές από κράτη-μέλη. Δεν χρειάζονται πλέον αυτή η προσωρινή ε, συνολική έλεγχη και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το, ε, πρέπει να μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τα αγαθά. Βρισκόμαστε στη διαδικασία αναθεώρησης των ε, κεντρικών ευρωπαϊκών συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και την εξασφάλιση της δηλαδοτικότητάς τους. Αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που θα μας βοηθήσει στην εξασφάλιση, στην ασφάλεια της, ε, του χώρου Σέγγεν. Αλλά Θέλω να επανέλθω στο ζήτημα ε, του, ε, του, στο εξή ότι το, το σύστημα ασύλου με τα προβλήματα που ε, αντιμετωπίζει συνδέεται άμεσα με το χώρο Σέγγεν και τα αντίστοιχα τα εκεί προβλήματα. Θέλω να πω λοιπόν ότι το, το συντομότερο δυνατό πρέπει να περάσουμε από αυτή τη χαόδη, χαοτική κατάσταση και να περάσουμε σε, μια καλά, σε ένα καλά οργανωμένο σύστημα μετανάστευσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και για τον χώρο Σέγγεν. Υπάρχουν στοιχεία ενδείξεις έχουμε ακούσει ε, εμπειρογνώμονες που μας ε, το έχουν επισημάνει αυτό με απόλυτη σαφήνεια. Το κάνω και εγώ λοιπόν. Χρειαζόμαστε το χώρο Σέγγεν και χρειαζόμαστε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Το συντομότερο δυνατό. Και να ξαναστραφώ στον κύριο Κοέλιο και να τον ξαναευχαριστήσω για το εξαιρετικό του έργο, για την εξαιρετική έκθεση και να του πω ότι προσβλέπω και στη συνέχιση της εξαιρετικής μας συνεργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Σεσίλια. Κάρλος, θέλεις να κάνεις κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Γκυγιόμ και την κυρία Βίξ για τα λόγια τους. Συμφωνώ με την άποψή σας για το ότι είναι απαραίτητο να εστιαστούμε στα πιο σημαντικά και να μην ξεχνούμε όμως και τα υπόλοιπα. Γιατί όπως ξέρει καλά η κυρία Βίξτρον και μας το είπε υπάρχουν προβλήματα σε επίπεδο Συμβουλίου. Ήδη είναι λυμμένη η απόφαση και μιλάω για το σύστημα ασύλου, για τη νέα υπηρεσία ασύλου, αλλά υπάρχει καθυστέρηση ανταπόκρισης όσον αφορά τα προβλήματα. Χρειάζεται παρέμβαση εκεί που χρειάζεται. Έτσι όμως διακυβεύεται η τύχη του Σέκεν. Θα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα του Σέγγεν για να μην ξεχάσουμε τον σκοπό του και να επίσης να λάβουμε υπόψη τις παράπλευρες συνέπειες για το έργο μας. Όμως δεν απόκειται σε εμά να αποφασίσουμε. Τα κράτη-μέλη πρέπει να αποφασίσουν και να μην συγχαίουν το Σέγγεν με άλλα. Αν θέλουν το Σέγγεν να εξυπηρετεί τους πολίτες, θα πρέπει να δωρακίσουμε την ελεύθερη διακίνηση. πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Και αυτό απασχολεί και την ε, Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι ως αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι υπάρχει συνένεση γύρω από αυτό το ζήτημα δεν μας εκπλήσει βέβαια αυτό και χαίρομαι για την μελλοντική συνεργασία με την κυρία Κιγιόμ, την κυρία Βίξτον και όλους τους άλλους σκιώδες προκειμένου να καταλήξουμε στην ευρύτερη δυνατή κοινή θέση, όπως είπα και εισηγητικά. Θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο αυτό πρέπει να στείλει ένα σαφέστατο μήνυμα στο Συμβούλιο και όσο μεγαλύτερη συνένεση υπάρξει εδώ, τόσο δυνατότερη θα είναι η φωνή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάρλος για την εξαιρετική αυτή η έκθεση και συμφωνούμε για το μήνυμα που μεταδίδεις. Ε, λοιπόν, προθεσμή είναι 14 Μαρτίου για τις τροπολογίες. Μία το μεσημέρι. Θα ήταν και το τελευταίο θέμα στη σημερινή σχεδιάταξη. διάταξη. Η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 12 Μαρτίου, 7 με 9 στο Στρασβούργο, ναι, ναι. Και 19 Μαρτίου, 5 ε, και 6.30 και μετά 20 Μαρτίου, πρωί και απόγευμα. Σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Α! Και σβήνει το μικρόφωνο του Πρόεδρου. Ναι, ναι, χρόνια πολλά στις ε, γυναίκες λόγω της ημέρας.